friends, Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με 11 λεπτά καθυστέρηση. Καταρχήν, να σας ενημερώσω ότι έχουμε μια μικρή αλλαγή στην μέση διάταξη, το σημείο 4 ακρόαση του οριστέντος διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα σημεία 5 και 6 συνεδρίαση αξιολόγηση από του συντονιστέ μετά την ακρόαση του οριστέντος διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Επαγγελματική Κατάρτιση ακυρώνονται. Και το 6. Η ψηφοφορία για το 11 δημοσιονομικοί κανόνε που εφαρμόζονται στο Γενικό προπολογισμό της Ένωσης αναβάλλεται. Θα λάβει η χώρα κάτι διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο να θέσουμε ερωτήματα και να ακούσουμε τους επιτρόπους, παρόλο που βέβαια και αυτοί έχουν τους χρονικούς τους περιορισμούς. Αύριο επίσης θα ξεκινήσουμε στις 9.30 και όχι στις 9. Μπορείτε να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω λοιπόν το πρωί. Κατά τα άλλα μπορούμε να δεχτούμε την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Ναι. Όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες εκτός φινλανδικών, κροατικών και ιρλανδικών. Να καλωσορίσω επίσης 28 εκπαιδευόμενους της Γενικής Διεύθυνσης μετάφρασης τραντ που είναι παρόντες ως ακροατές. Καλώς ήρθατε, θερμά σας καλωσορίζουμε. Για να δείτε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Οι περισσότεροι στην πράξη μιλούν κακά αγγλικά. Ελπίζω εσείς να μας βοηθήσετε λιγάκι κάποια στιγμή στην καριέρα σας. Περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων ως τμήμα του διαρθρωμένου διαλόγου με τον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσκης και την Επίτροπο την κυρία Μαριάν Τάισεν. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκης. Παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου και να ε, εξετάσουμε την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας κομισιών για φέτος. Ε, το πρόγραμμα εργασίας του 2007 ήταν φιλόδοξο προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική σύγκληση και η κοινωνική διάσταση Ευρώπης. Βασική μας ε, δέσμευση ήταν το Ευρωπαϊκή Χάρτα ε, κοινωνικών δικαιωμάτων και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Μια δημόσια διαβούλευση μας έδειξε το δρόμο και πήραμε υπόψη και την έκθεση του περασμένου Ιανουαρίου. Η Επιτροπός Τάισεν και εγώ ίδιος την περασμένη εβδομάδα ε, υποβάλαμε το νομοθέτημα μόλις υιοθετήθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Το παρουσιάσαμε μάλλον. Ε, επίσης συνοδεύεται από διάφορε πρωτοβουλίες που αποτελούν τμήμα του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι ένα συγκεκριμένο βήμα που δείχνει ότι η κοινωνική διάσταση δεν είναι κάτι το αφηρημένο για μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια, είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει τις ζωές όλων των πολιτών. Με την υλοποίηση της υπόσχεσης για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μας. Η Επιτρόπος κυρία Τάισεν θα μας ε, παρουσιάσει με περισσότερες λεπτομέρειες τις προτεραιότητες που καταγράφηκαν στην κοινή δήλωση. Να πω όμως ε, να σχολιάσω αυτό που, σχολιά, που υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ. Ε, δύο θέματα για τα οποία θα χρειαστούμε τη δημόσια διαβούλευση. Πρώτον, πρόσβαση, ε, μάλλον πρωτοβουλία για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Κοινωνική προστασία που καλύπτει ε, εργαζόμενους ε, σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας αποτελεί ένα αντικείμενο, αποτέλεσε αντικείμενο και στο παρελθόν. Η επίσημη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους έληξε την περασμένη εβδομάδα. Κοινωνική διαβούλευση που αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλες τις μορφές εργασίας, ιδιαίτερα τους ανέργους, οι οποίοι θέλουμε να έχουν ίση πρόσβαση. Με αυτή την πρωτοβουλία ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας να υιοθετηθεί μια οδηγία πλαίσιο που να αφορά όλους τους τύπους εργασίας. Δεύτερον, ε, θέλουμε να κάνουμε βήματα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τον τύπο σήμασή τους να χαίρουν των ίδιων προνομίων. Πολλοί εργαζόμενοι, για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν γραπτή γνωστοποίηση των όρων εργασίας γέρος. Μεταξύ αυτών η οικιακή βοηθή και ε, αυτοί που ε, εργάζονται σε βάρδιες. Η συνθήκη μας ε, απαιτεί από μας ε, να διαβουλευτούμε με τους κοινωνικούς εταίρους στα περισσότερα από αυτά τα θέματα. Η διαβούλευση αυτή καλύπτει ε, πιο ευρείες ζώνες και αυτό το λόγο ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση και όχι μόνο διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Επίτροπος Τάισεν και εγώ ο ίδιος αναμένουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για αυτές τις πρωτοβουλίες του κοινωνικού πυλώνα έτσι ώστε πραγματικά να κάνουμε μια σημαντική τη διαφορά στην ζωή των πολιτών μας. Ο διαθετημένος διάλογος έχει σχέση και με τα μελλοντικά σχέδια πρόγραμμα εργασίας κομισιών. Ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, ε, και η Κομισιόν ε, υιοθέτησαν το ε, νόμο για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και σκοπεύουμε να αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν θα λάβει δράση, θα λάβει πρώτον στην εφαρμογή της ισχύωσης νομοθεσίας ιδιαίτερα με το input των κοινωνικών εταίρων θα δούμε πού υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του κοινωνικού κεκτημένου και θα αποφασίσει τη δράση πρέπει να αναλυθεί. Δεύτερον, θα παρακολουθήσουμε καλύτερα την πρόοδο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα προτείνουμε ένα καινούριο κοινωνικό βαθμονόμιο, όπως ακριβώς ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, να επαναλάβω ότι ο βασικός μας στόχος είναι η κοινωνική και η κοινωνική σύγκληση να πηγαίνουν παράλληλα. Επίσης, Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, δημογραφικές αλλαγές, ε, η παγκοσμιοποίηση και άλλα. Το έγγραφο σκέψη για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης ακριβώς λαμβάνει υπόψη όλα αυτά και παρουσιάζει τις ε, δυνατότητες ε, πολιτικής για το μέλλον. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει βάση της συζήτησης για τους επόμενους μήνες και θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε την πολιτική μας για την κοινωνική διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναμένω ε, τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Και τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο, την κυρία Τάισεν. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, Βάλντις, συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μια κοινωνικότερη Ευρώπη είναι μια κοινή μας επιδίωξη, ημών των συνομοθετών. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων δίνει έμφαση στην κοινωνική διάσταση στην κοινωνισματική Ένωση. Έχουμε σχεδιάσει τον πυλώνα ω έναν τελικό στόχο για να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση και να έχουμε καλύτερε εργασιακέ και συνθήκες, και συνθήκες διαβίωση στην Ευρώπη. στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν η σωστή υλοποίηση αυτού του πυλώνα να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στους Ευρωπαίους πολίτες και να ανοίξει το δρόμο μας προς την πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα υπόψη ως πρωτοβουλίε για τους εργαζομένους και την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, των χρόνων εργασίας, όπως τα ανέπτυξε ο Βάλντης. Εγώ να αναφέρω την νομοθετική πρόταση που υποβάλαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον Πιλώνα. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προωθήσει μέτρα για τη βελτίωση τη εξισορρόπηση επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Ακολουθούμε μια ευρύτερη προσέγγιση για να δούμε την ε, μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στην ε, αγορά εργασία. Λαμβάνουμε υπόψη τι εξελίξει στην κοινωνία την τελευταία δεκαετία και ενθαρρύνουμε την καλύτερη κατανομή των ευθυνών ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών για τη φροντίδα, της ε, υπηρεσίας φροντίδας. Εδώ έχουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για να βελτιωθεί το πλαίσιο στους τομείς ε, της άδειας που έχουν σχέση με τον οικογενειακό βίο και την, τον ευελιξία στο χρόνο εργασίας. Επίσης συμπληρωματικά μέτρα, δικουρικά μέτρα για να μπορέσουμε να έχουμε φροντίδα σε καλή τιμή στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι και να δίνονται κίνητρα και στους ε, εργαζομένους, ώστε να είναι ικανοποιητική η προσφορά κινήτρων και στους διογόνεις. Αυτά καταγράφονται και στην κοινή μας δήλωση. Να ξεκινήσω με την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα ζητήματα αυτά για τους πολίτες ε, στις ε, εθνικές συζητήσεις και στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή. Και για να έχουν οι πολίτες μας μεγαλύτερη κινητικότητα και να κυκλοφορούν στην Ένωση, θα πρέπει να θεωρούν ότι οι συνθήκες είναι δίκαιες, ότι προσφέρονται ευκαιρίε σε όλους. Και ότι δεν μπορούμε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αντιπαραθέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Το πρώτο στοιχείο της ε, κινητικότητας είναι ακριβώ η ε, αναθεώρηση τη οδηγία για την απόσπαση. Και να ευχαριστήσω εδώ τι εισηγήτριε, την κυρία Γιονκέριου και την κυρία Μωρέν Σαρτιέ, για όλη του τη δουλειά και τι άοκνε προσπάθειέ του για αυτό το θέμα. Ε, καλωσορίζω το σχέδιο έκθεσή σα. Πιστεύω ότι έχετε πετύχει ένα πολύ καλό σημείο ισορροπία. Ελιζαμπέτ, δεν σε είχα δει, με συγχωρείς. Ε, πιστεύω ότι και οι δυο σα μαζί πετύχατε ένα σωστό σημείο ισορροπίας ε, με τις κοινωνικές προδιαγραφές για την δικαιοσύνη, ενώ έρονται τα ε, εμπόδια για τις εταιρείε που θέλουν να προάγουν την ε, κινητικότητα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο τον Ιούνιο ήδη επί της Προεδρίας αυτής. Το να πετύχουμε συμφωνία είναι περισσότερο ε, από ποτέ σημαντικό τώρα. Το περιμένουν οι πολίτες μας για την εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε πλέον να αφήνουμε κενά και παραθυράκια, διότι αυτό ακριβώς πυροδοτεί τις αντιρρήσεις εναντίον μας που προωθούν απλουστευμένες και δραστικέ λύσεις. Ελπίζω να πετύχουμε λοιπόν τη συμφωνία για το θέμα αυτό πολύ γρήγορα για μια Ευρώπη κοινωνικότερη και για να επικεντρωθούμε στις πτυχέ που μας ενώνουν, μα φέρνουν πιο κοντά και όχι αυτές που μας οδηγούν σε διαφωνίε και μας χωρίζουν. Το δεύτερο μέρο του, του πακέτου για τις για την κινητικότητα έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση. Στις 23 Μαρτίου υπέβαλα την πρότασή μας ε, σε σχέση με τους κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση και τον συντονισμό. Ε, εδώ έχουμε μια εξισορροπημένη πρόταση για να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύουμε τις εθνικές αρχές που θα μπορούν να καταπολεμήσουν την κατάχρηση ή την απάτη. Είναι επίκαιρη η έλευση αυτή της ε, οδηγία για να είναι σαφείς οι συμβολές και ε, ξεκάθαρα τα δικαιώματα και να υπάρχει και μια σωστή κατανομή των ευθυνών μεταξύ των χωρών. Όπω προείπα, η πρόταση δεν τροποποιεί ισχύοντε κανόνε για την ε, εξαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η χώρα της εργασίας των γονέων παραμένει ε, υπεύθυνη για τα επιδόματα των παιδιών. Και τα ποσά αυτά μπορούν να προσαρμοστούν εφόσον το παιδί διαμένει κατοικεί αλλού. Τα επιδόματα για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί λοιπόν να εξαθούν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Αυτή η πρόταση, όπω ξέρετε, είναι μία από τι νομοθετικέ προτεραιότητε που αναφέρεται και στην κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων και καλωσορίζω τον διορισμό του εισηγητού Μπαλά και ελπίζω ότι μαζί θα κινηθούμε σωστά για να πετύχουμε και την περάτωση την ολοκλήρωση του θέματος αυτού. Τώρα, η προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα. Εδώ ήθελα να προτείνω νέα όρια για την επιτρεπόμενη έκθεση όσο δυνατόν συντομότερα. Ε, για την κάθε ουσία υπάρχει μια λεπτομερής αξιολόγηση του κόστους και της ωφελίας που ε, επιφέρουν και γι' αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε σε τμήματα με τις χημικές ουσίες για τις οποίες πληροφορίες διαθέτουμε σε αυτονία. Ήδη έχουμε υποβάλει τα δύο πρώτα και αυτές οι δύο προτάσεις επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλεπόταν στο πρόγραμμα το 2016, να ε, πετύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ελπίζω και εδώ να πετύχουμε συμφωνία και για το τρίτο τμήμα το μελετούμε αυτή τη στιγμή, ώστε καινούργια πρόταση να γίνει στις αρχές του 2018 με επιπλέον ουσίες που έχει ήδη σχεδιαστεί ε, ως δουλειά. Εδώ εκτιμώ τις προσπάθειες των συναδέλφων που μελετούν αυτά τα θέματα και όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφκης, ε, Ανυπομονώ για τη συνεργασία μα για τι νέε αυτέ πρωτοβουλίε που αφορούν τον πυλόν των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα τονίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι τώρα που όλε οι προτάσει ε, βρίσκονται μπροστά μα επιτάπητο και είναι σημαντικό να πετύχουμε ε, ένα σημείο σύγκληση και συμφωνία χωρί καθυστέρηση. Για κάθε νέο νομοθέτημα ε, θα πρέπει με κάθε μάλλον νέο νομοθέτημα, αποδεικνύουμε στου πολίτε μα ότι η κοινωνική Ευρώπη είναι πραγματικότητα. Η Ευρώπη μπορεί όντω να φέρει μια διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Με καλύτερη νομοθεσία και κυρίω προτείνοντα ε, δείκτε συγκριτική αξιολόγηση και δείχνοντα ποια είναι τα αποτελέσματα των κοινωνικών μα προσπαθειών τώρα. Ε, είμαι πάντα στη διαθέσή σα για να συζητήσουμε και αναμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Τάισεν. Και τώρα ο κύριος Μπέκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Πολύ θετικά αντιμετωπίζω την παρουσίαση που κάνετε την προηγούμενη εβδομάδα ίση πρόσβαση στην αγορά εργασία με δίκαιες συνθήκε εργασία και επαρκείς και βιώσιμες ε, ρυθμίσεις κοινωνικής προστασίας είναι στο επίκεντρο της ε, ανακοίνωση αυτής. Και κάτι άλλο που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι θεωρείται ότι η βάση για όλα που επιδιώκουμε τώρα είναι η πολιτική για μια κοινωνική αγορά. Επίσης, Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχουν νέες προτάσεις για νέα μέτρα, για την εξορρόπηση προσωπικού και επαγγελματικού βίου, που είναι η πεμπτουσία των προσπαθειών που κάνουν εκατομμύρια συμπολιτών μας. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Ε, δυστυχώς, για να επιτύχουμε περισσότερη απασχόληση δεν πρέπει να εργαζόμεθα εν κενό. Πρέπει να, να αυξάνουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων μας. Η αγορά γίνεται όλο και πιο ψηφιακή. Οι τεχνολογίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αλλά πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δεξιότητες για αυτές. Καλό την Επιτροπή να μην ξεχάσει επίσης ε, τη σημασία της διαβίου κατάρτισης. Αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, σαφές. Αλλά βοηθάει πολύ το ότι το προβάλλετε τόσο πολύ. Παρακαλώ συνεχίστε. Για να μπορούν να επανέλθουν και οι μεγαλύτερες ηλικία εργαζόμενοι στην αγορά εργασία και άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Να διευκρινίσω κάτι. Θεωρώ ότι εσείς ε, ως Επιτροπή καταλαβαίνετε σαφώς πόσο σημαντικές είναι οι εθνικές αρμοδιότητες για να νομοθετούν για τα θέματα αυτά. Είναι λοιπόν πολύ υπεύθυνη η προσέγγιση σας. Γιατί τονίζετε σαφώς ότι και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή είναι πολύ ευφυής, πολύ επικοδομητική στάση και θα βοηθήσει την ανάπτυξη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Η κυρία Γιονγκέριους. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, την παρουσίαση των ε, προθέσεών σας. Είπε κάτι ο κύριος Ντομπρόφσκης ότι θέλουμε να κάνουμε διαφορά στη ζωή και την καθημερινότητα των ε, συμπολιτών μας, των απλών ανθρώπων στην Ευρώπη. Όμως, σκεπτόμενοι πώς θα τα επιτύχουμε αυτά, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσω κάπως διαφορετικά τις προτάσεις της προηγουμένης εβδομάδας. Καταρχάς, σας συγχαίρω για την εργασία σας, για την ε, απόσπαση των εργαζομένων, την οδηγία γι' αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι ο συνάδελφος Μπάλας εργάζεται επικοδομητικά για τα θέματα της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και ότι και οι καρκινογόνες ουσίες προχωρούν. Αλλά βλέποντας το πακέτο που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τότε είμαι λίγο πιο επικριτική. Βεβαίως σημαντικό ότι έχουμε αυτή την πρόταση για συνδυασμό ιδιωτικού βίου και εργασίας. Αλλά δεν έχουμε προτάσεις για την άδεια μητρότητας, δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο. Και δεύτερον, αν θέλουμε δίκαια και ισότιμη κινητικότητα των εργαζομένων, πρέπει πράγματι να αλλάξουν κανόνες. Αλλά, αλλά, θέλουμε να υπάρχει και διασυνοριακή ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας και να προωθηθεί και η Κάρτα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλισης. Και θέλουμε να γίνουν περισσότερα για τα παιδιά, για την παιδική ανέχεια. Αλλά δεν έχουν γίνει συγκεκριμένε προτάσεις ακόμη. Δεν υπάρχουν στο πακέτο. Και τέλος, και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό που αναφέρω, είναι ότι ναι μεν και επειδή είμαι συνδικαλίστρια εκτιμώ ιδιαίτερα τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τις οδηγίες αυτές, τις δύο αυτές οδηγίες. Αλλά πραγματικά πιστεύω επίσης ότι θα ήταν σκόπιμο να καταστήσει σαφές η Κομισιόν προς τους κοινωνικούς εταίρους ότι εάν η διαβούλευση για την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση για όλους τους εργαζόμενους με κάθε τύπο εργασίας. Εάν δεν καταλήξει σε προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή θα υποβάλει παρόλα αυτά προτάσεις. Γιατί αλλιώς φοβάμαι. ότι θα κάνουμε διαβουλεύσεις για τις διαβουλεύσεις. και δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και εργαζομένων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τους επιτρόπους που είναι εδώ παρόντες σήμερα. Το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν που μας παρουσίασαν είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε πολύ υψηλές κοινωνικές ε, προδιαγραφές και δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αναγκαστικά και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις ή να παρεύουμε εκεί που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γιατί ξέρετε ότι οι κοινωνικοί παράγοντε ε, παίζουν ρόλο στο κόστο παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε αυτό το τόσο φιλόδοξο πακέτο και για την ομάδα μου αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να προσφέρουν ε, προστιθέμενη αξία στους πολίτες αυτές τις πρωτοβουλίες που δεν θα την είχαν χωρίς την παρουσία και παρεμβολή της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη όμως δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Η ανταγωνιστικότητα και η επιβίωση των μικρομεσαίων δεν θα πρέπει να θυγούν. Συγκεκριμένες ερωτήσεις για λεπτομέρειες τώρα. Έχετε λοιπόν σχέδια σε αυτή τη φάση για την εφαρμογή νομοθετημάτων που ήδη υπάρχουν, όπως για την ε, ε, οδηγία για την ε, διάρκεια, τα ωράρια της εργασίας. Και επίσης, τονίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στις πρωτοβουλίες και στα αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί. Και το θέμα είναι και να εφαρμόζετε καλύτερα η νομοθεσία, να αποδώσετε περισσότερο βάρος σε αυτό. Για παράδειγμα, να συμμετάσχουν περισσότερο κοινωνικοί εταίροι και να έχουμε και μελέτες ε, συνέχεια, ούτω ώστε να υποβάλλετε τα αποτελέσματα και στην Επιτροπή για τον έλεγχο των ρυθμίσεων, για να αποφευχθούν λάθη και κάτι άλλο. Τι κάνει η ίδια Κομισιόν για να ε, ενημερώσει για τους ε, μακροοικονομικούς δείκτες, τους ε, μακροοικονομικούς σταθεροποιητές. Να ενημερωθούν λοιπόν, γιατί δεν ενημερώνουν αρκετά οι εθνικοί φορείς για το τι μπορεί να κάνει για αυτούς η Ένωση, τους πολίτες τους. Ευχαριστώ ε, ο κύριος Καλβά Σαμπό. Κάλβε Τσάμπο Καλώς ήρθατε ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επιτροπή, θα απευθυνθώ καταρχήν στα Ισπανικά στον κύριο Αντιπρόεδρο. Με ακούει? Να δούμε να προλάβει να βάλει λίγο τα ακουστικά του. Ωραία. Με ακούτε κύριε Ντομπρόσκης. Ωραία. τρεις τύπους ορισμού της κοινωνικής Ευρώπης έχετε προβάλει. Αναμφίβολα η, η κοινωνική Ευρώπη σήμερα είναι ε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ε, Ευρώπης και των πολιτών της. Και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αν ήμασταν μόνο μια αγορά με εμπορικέ συμφωνίες ή ε, ε, τότε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν το κοινωνικό κομμάτι να αφαιθεί στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας πω το εξής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την επικουρικότητα. Η επικουρικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αποκέντρωση. Όμως αυτό για το οποίο μιλάμε είναι τα βασικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Άλλο αυτό και άλλο η εφαρμογή αυτού να πρέπει να γίνεται κοντά στους πολίτες, δηλαδή με αποκέντρωση και επικορικότητα. Θα πρέπει να ρωτηθούμε, θα είναι καλύτερη η κοινωνική ζωή των πολιτών μας, αν είναι σε μια Ευρω... Ε, ενωμένη Ευρώπη. Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αν οι πολίτες μας βρίσκονται σε μια ενωμένη Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και ε, οικονομική αλληλεγγύη για τον κοινωνικό τομέα. Αυτά. Και να τελειώσω στα γαλλικά για την κυρία Τάισεν, για να με ακούσετε χωρίς διερμηνία. Πολύ καλά όλα αυτά που προτείνετε, αλλά ε, σκεφτείτε δύο πράγματα για το μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος στην κοινωνική Ευρώπη και με αλληλεγγύη να μην μιλήσουμε για την φτώχεια και την ακραία φτώχεια που θα πρέπει να διαγραφούν από την Ευρώπη, να εξαφανιστούν. Η Κομισιόν θα, πάρει, θα λάβει μέτρα γι' αυτό. Δεύτερον, δεν, υπάρχει, δεν θα βελτιώσουμε την κοινωνική Ευρώπη αν δεν καταπολεμήσουμε, σε συνεργασία εσείς με τον κύριο Ντομπρόφσκης, με την οικονομική και την κοινωνική πολιτική, την αύξηση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στην κυρία Ρενιακάρη. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Ο κοινωνικός πυλώνας ε, βρίσκεται στο επίκεντρο των αισιών μας εδώ και καιρό. Κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε παντού στην Ευρώπη. Αυτά που προτείνατε την περασμένη εβδομάδα βασίζονται στις 20 αρχές και το κοινωνικό βαθμολόγιο. Όμως, ε, και ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή υφίσταται ένα σύστημα ελέγχου της οικονομίας και των οικονομικών στοιχείων του κάθε κράτους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πώς θεωρεί ο Κομισιόν ότι συνδέεται το κοινωνικό βαθμολόγιο με τις ε, συστάσεις περί Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι, κοινωνικές, ε, οι κοινωνικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να βρεθούν στο επίπεδο των οικονομικών απαιτήσεων. Δεύτερον, η, ψηφιακή οικονομία. Ε, έχετε προτείνει μια στρατηγική για αυτήν. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι εκεί στην ψηφιακή οικονομία οι εργαζόμενοι θα χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Ε, ή στην οικονομία με τις διάφορες πλατφόρμες όπως η Uber και άλλες. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, περί κοινωνικού πυλώνα. Τα, θε, τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα είναι απόλυτα σημαντικά. Πώς όμως συνδέονται με το πακέτο περικινητικότητας. Εντοπίσαμε τα κενά τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνική κοινωνικής ασφάλισης ε, και, και πώς συνδέεται αυτή με την κοινωνική βοήθεια και συνδρομή. Για παράδειγμα, Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι αναγκάζονται να ε, έχουν μείνει άστεγοι ή θα ε, πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα στην οποία διαμένουν επειδή δεν εγκαλύπτονται κοινωνικά πώς, ε, ε, λειτουργεί ο συντονισμός μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων όταν οι εργαζόμενοι μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν να τα έχετε εντοπίσει. Δεύτερον, η σχέση ανάμεσα στις επαγγελματικές ικανότητες και την κυκλική οικονομία και την πράσινη οικονομία. Ποιες είναι, πώς διαρθρώνεται το έργο, οι εργασίες της Κομισιόν έτσι ώστε η ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων να συνδεθεί με την κυκλική οικονομία. Προφανώς ε, κάποιοι έχουν βαρεθεί εκεί πίσω γιατί έχω ε, μακρηγορήσει υπερβολικά. Ευχαριστώ, η Λάουρα Αγκία δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσω το λόγο στον Ντομινίκ Μαρτά. Ο διαστατημένος διάλογος ε, που λαμβάνει η χώρα ετησίως ε, μας καλεί να σχολιάσουμε το πρόγραμμα που μας προτείνει η Κομισιόν κάθε φορά και ε, πάντοτε ε, υπό πομπόδιες τίτλους. Το 2015 το πρόγραμμα της Κομισιόν είχε τίτλο «Μια καινούργια αρχή», «Μια καινούργια όθηση», συγγνώμη, το 16 έχει περάσει ο χρόνος της συμβατικής διαχείρισης και φέτος ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες μιας Ευρώπης που προστατεύει και που δίδει τα μέσα δράσης. Το, η ορολογία που χρησιμοποιεί η Κομισιόν βλέπω εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Εξού και δυσκολευόμαστε να υποβάλουμε προτάσεις και να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα της Κομισιόν γιατί το κείμενο αυτό ε, έρχεται να ε, ε, ενισχύσει το ρόλο της Κομισιόν και τις παρεμβάσεις της σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή Απασχόλησης, ακόμα και όταν η Επιτροπή Απασχόλησης έχει προτάσει να κάνει, η απάντηση συνήθως είναι ίδια. Ε, άρνηση. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ε, Κομισιόν, κυρία Επιτροπέ, και πάλι πρόκειται για ένα ασαφές κείμενο, γεμάτο με καλές προθέσεις, χωρίς όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Είτε σε ό,τι αφορά τις δάσεις, είτε σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ο προγραμματισμός δεν είναι σαφής. Από ό,τι φαίνεται ο στόχος σας είναι, βλέπετε, οπότε ε, βλέπετε υπάρχουν διαφωνίες ήδη στην αίθουσα. Κάθε φορά έχουμε τις ίδιες απορίες, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια αιτήματα. Σε ό,τι αφορά τη δική μας συνεισφορά. Ε, όλες σας οι όλες αυτές οι δράσεις είναι παρεμβάσεις της Κομισιόν στο έργο των κρατών μελών. Πάντοτε μπλέκεστε όλο και περισσότερο στα, στις δραστηριότητες της αρμόδιας των κρατών μελών, είτε ζητώντας τους καινούριε πολιτικές, είτε ζητάτε στα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσουν το πώς εφαρμόζονται ε, τα προγράμματά σας. Ε, ίδιες διαπιστώσεις και προφανώς η ίδια κρίση κάθε φορά από μέρους μας. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Μαρτά. Πριν συνεχίσουμε με τον κατάλογο των αγορητών, θα δώσω το λόγο στους επιτρόπους μας για να απαντήσουν. Πρώτος ο κύριος Ντομπρόφσκης και μετά κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές αρκετές παρατηρήσεις, οπότε θα προσπαθήσω να τις σχολιάσω εντάχει. Για τον κύριο Μπέκερ πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, για τα θέματα που αναφέρατε και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες, το skilling. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία όντως θέλουμε να δώσουμε έμφαση με την ε, το κατάλογο προτεραιοτήτων για τις δεξιότητες. Διότι οι μέθοδοι εργασίας αλλάζουν, οπότε αλλάζουν και, οι δεξιότητες που απαιτούνται. Για συγκεκριμένου λόγου, λόγου χάρη μιλήσουμε για την ψηφιακή οικονομία, για παραδείγματα. Σαφώ αυτέ είναι ε, από τις πρώτε μας προτεραιότητε. Οι δεξιότητε των εργαζομένων να παραμείνουν ε, ανάλογες με τις απαιτήσει της αγοράς εργασίας και να υπάρχει πρόσβαση σε ποιοτικέ θέσει εργασία. Και για τις ερωτήσεις σας, κυρία Γιονγκέριους, Δείξατε πολλά σημεία για την δίκαιη, την ισότιμη κινητικότητα. Μας απασχολεί αυτό. Το δείξαμε και με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και με άλλους τομείς για το θέμα της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το θέσατε για το θέμα της ε, κοινωνικής ασφάλισης και της σχετικής οδηγίας, όντως ξεκινούν τώρα διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία από παιδευτέρων. Αυτό φάνηκε και με την πρωτοβουλία μας για την εξισορρόπηση επαγγελματικού οικογενειακού βίου και την γονική άδεια, όπου είχαμε ακριβώς τέτοιου είδου συνθήκε. Τώρα για τα ερωτήματα για την οδηγία χρόνου εργασία. για την ώρα στο επίπεδο της ερμηνείας για να δούμε την ομολογία και τις αποφάσεις του δικαστηρίου σε αυτό το επίπεδο και τα κάτι μελη να έχουν περισσότερες ε, συγκεκριμένες οδηγίες για τους εργοδότες και να δουν πώς οι βασικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτό το τομέα. Παρόμοια και για την ερώτησή σας για την ε, καλύτερη νομοθεσία. Ακολουθούμε προφανώς αυτές τις αρχές Και αυτό μα απασχολεί και στον πέδο τη υλοποίηση. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αποτιμούμε κατά πόσον υπάρχουν κενά ή ελλείψει στην υλοποίηση και προσπαθούμε να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση για να αντιμετωπίσουμε ακριβώ την ύπαρξη κενών. Μετά, συγκεκριμένη ερώτηση τέθηκε για την οικονομική στήριξη της κοινωνικής διάστασης. Πρώτα απ' όλα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς και επίσης προσφέρουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια σε μια νέα στόχευση για να καλύψουν ακριβώς κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες της κοινωνικής κατάστασης. Ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και τώρα στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και στις συζητήσεις για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις και συγκεκριμένε κατευθυντήριες γραμμές για να μπορούμε να δούμε πώς θα καλυφθεί ακριβώς η κοινωνική διάσταση. Και βάσει της συνθήκης, αυτά τα θέματα παραμένουν πρωταρχικώς ευθύνη των κρατών μελών ούτως ή άλλως. Αναφέρατε επίσης το θέμα της μείωσης των ανισοτήτων, της άμπληξης των ανισοτήτων. Εδώ είναι ένα από τα βασικά σημεία προτεραιότητα ε, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όταν μιλάμε για τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή και την ετήσια έκθεση, ακριβώ υπογραμμίσαμε την ανάγκη να αμπλυνθούν οι ανισότητε. Αυτό έρχεται να ε, σχετιστεί και με την επόμενη ερώτηση για το βαθμολόγιο. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επικεντρωθήκαμε επανειλημμένο στο γεγονό ότι οι οικονομικές και κοινωνικέ υποθέσει πρέπει να συμβαδίζουν. Το κοινωνικό λοιπόν βαθμολόγιο θα μα δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να αποτεμήσουμε ευκολότερα την πρόοδο στα κατημέλη, ώστε να απηχείται και στι αναχώρασει τάση, όπω είπα προηγουμένω με στόχο να μειωθούν οι ανισότητε λόγω του εισοδήματο. για την ψηφιακή οικονομία, τις πλατφόρμες της ψηφιακής οικονομίας. Αυτή είναι μια από τις βασικές μας πρωτοβουλίες τώρα. Πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους ασχέτως της μορφής απασχόλησης όπου απασχολούνται. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές εργασίας πλέον και πρέπει να είμαστε στο ρυθμό των εξελίξεων. Για την ερώτηση που τέθηκε για την κοινωνική ατζέντα και τις πράσινες θέσεις εργασίας και την κυκλική οικονομία, αλλά και τον κατάλογο προτεραιοτήτων μας ε, για τις δεξιότητες σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία και τις πράσινες θέσεις εργασίας. Σύντομα, προς το τέλος του μήνα, θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τις πράσινες δουλειές. Το επεξεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους. και θα υπάρξει μια πολύ ε, χειροπιαστή εξακολούθηση πρόθεση του θέματο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πάψω εδώ προς τη Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Τάισεν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, Εφόσον έχω δυνατότητα θα μιλήσω τη γλώσσα μου. σας αφήνω λίγο χρόνο να διαβάλλετε τα ακουστικά σας. Κύριε Μπέκερ, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τη θετική σας ε, αποτίμηση. Και εμείς εργαστήκαμε πολύ, αλλά και εσείς, γιατί υποβλήθηκε μια θαυμάσια έκθεση κατά την ε, διάρκεια Εκπόνηση των θέσεών μας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας τη συμβολή και χαίρομαι που μπορούμε από κοινού να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόοδου, υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τονίσατε πόσο σημαντική είναι η σωστή κατανομή ε, αρμοδιοτήτων. Βεβαίως. Συγγνώμη, εννοώ μάλλον τις δεξιότητες. Τις δεξιότητες πρέπει να προωθήσουμε. Είναι το πρώτο σημείο. Ε, οι δεξιότητες θα επιτρέψουν να ε, τα πάνε καλύτερα ε, οι περισσότεροι για να υπάρχει ε, ίση δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσω της διαβίου κατάρτισης και φυσικά μέσω και των σωστών μέτρων κοινωνικής προστασίας. Να ευχαριστήσω και όσους αναφέρθηκαν στην διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για μας ε, είναι αναμφίβολα ένα από τα βασικά στοιχεία της όλης προσπάθειας. Ιδιαίτερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και νομοθετικά. Πάντα όταν ε, συζητάμε για νομοθετήματα, συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο γιατί μας επιβάλλεται από τις συνθήκες, αλλά γιατί μας βοηθάει αυτό. Ούτω ώστε οι προτάσεις, μας, να είναι καλύτερε. καλύτερες. Όταν γίνει σωστή και αποτελεσματική διαβούλευση, τότε έχουμε κάθε δυνατότητα κατόπιν να λάβουμε αποφάσεις που είναι απόλυτα εφαρμόσιμες με την κοινή μας προσπάθεια, λοιπόν, την κοινή μας καλή θέληση. Κυρία Γιονγκέρος, αναφερθήκατε στον συνδυασμό οικογενειακής και προσωπικής, ε, συγγνώμη, επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην προστασία των μητέρων, την άδεια μητρότητας. Ξέρετε ότι κάναμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση για να επιμηκυνθεί η άδεια μετρότητας, αλλά τελικά αποσύρθηκαν αυτές οι προτάσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποβάλουμε καλύτερες προτάσεις. Γιατί χρειάστηκε τελικά να αποσύρουμε την πρότασή μας, γιατί είχε μπλοκάρει στο Συμβούλιο από το 2008. Οπότε τελικά αποσύραμε την πρόταση για να επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Και βέβαια δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με την κατάσταση των μητέρων, αλλά και την κατάσταση των πατέρων και όλων όσων ασχολούνται με την ε, ε, φροντίδα, με την ανατροφή των παιδιών και το πώς θα μπορέσουν να συνδυάσουν αυτή τη φροντίδα με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ξέρουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη η άδεια μητρότητας ε, είναι πολύ μακρύτερη από αυτό που προβλέπει η οδηγία. Και διαπιστώσαμε επίσης ότι τίθενται και θέματα της προστασίας στον τόπο εργασία. Πρέπει να επιτρέπουμε στις γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να επιτυγχάνουν αυτό το συνδυασμό της ε, ε, προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε βεβαίως τις μητέρες, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει και πώς θα συμβάλλουν οι πατέρες. Είναι πολύ φιλόδοξη η πρόταση που, που προτιθέμεθα να κάνουμε και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Τώρα για την δίκαιη κινητικότητα, fair mobility. Ναι, κάναμε περισσότερα. Αλλά διαβάστε το έγγραφό μας ε, το ευρύτερο για την κοινωνική προστασία. Είναι το πρώτο έγγραφο συζήτησης που ξεκινήσαμε στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης. Και μία από τις λύσεις που προτείνουμε για συζήτηση, μία πρόταση δηλαδή, είναι ότι ναι μεν ε, θα μπορούσαμε να έχουμε Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Εργασίας, αναφερθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Όλα αυτά βεβαίως προωθούν περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά δεν συμμερίζονται όλοι, κυρία Γιονγκέριους, αυτή μας την προσέγγιση. Και όλα όσα μπορούμε να πούμε για το θέμα αυτό θα το βρείτε στην πράσινη βίβλιο λοιπόν για την κοινωνική Ευρώπη. Βεβαίως προτιθέμεθα να ε, έχουμε διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Αναφέρεστε επίσης στις ε, αυτόνομες συμφωνίες. Βεβαίως πρέπει να καθορίσουμε τις δυνατότητες λύσεων από την αρχή. Το είπε και ο Αντιπρόεδρος ε, Ντομπρόφσκης και ασχοληθήκαμε επίσης με το πώς πρέπει να γίνεται ένα γραπτό, μια γραπτή σύμβαση εργασίας. Βεβαίως να υπάρχει διαβούλευση. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης είναι η σημασία της ε, δυνατότητα παρέμβαση τη Κομισιόν. Η Κομισιόν θα πρέπει, αν δεν υπάρχει συμφωνία, να μπορεί να υποβάλει προτάσει. αν δεν υπάρχει συμφωνία δηλαδή με του κοινωνικού εταίρου. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν φυσικά οι κοινωνικοί εταίροι οι ίδιοι. Κυρία Τρεμπέσιους, αναφερθήκατε σε μια σειρά από νέα ζητήματα, καθώ και στην ανάγκη εφαρμογή τη νομοθεσία. Βεβαίω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ό,τι αποφασίζετε κατόπιν να εφαρμόζεται ιδίω όσον αφορά την προστασία στην αγορά, ε, στο, στον τόπο εργασία, από έκθεση για παράδειγμα σε καρκινογόνες ουσίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τρεμένη διάλογο επ' αυτού, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται άμεσα με αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε η εφαρμογή της νομοθεσίας να μας απασχολήσει και μας απασχολεί σε κάθε φάση. Διότι υπάρχουν νομοθετήματα που ήδη έχουμε εγκρίνει. Το θέμα είναι τώρα να εφαρμόζονται. Τώρα για τον πυλώνα γενικότερα. Κοιτάξτε, δεν ε, προτείνουμε νέα μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ένωση, όχι. Προτείνουμε απλώς κάποιες κοινέ αξίες, που ελπίζω τουλάχιστον να είναι κοινέ μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ούτω ώστε με βάση τις δικές μας αρμοδιότητες να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα μέσω της δράσης μας. Και αυτό προτίθεμεθα να κάνουμε. Βεβαίως ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος, διαθέσιμος, διατεθειμένος να αναλάβει τις ευθύνες που το αναλογούν. Κύριε ε, Καλβέτ Τσαμπόν, για τη φτώχεια και την ε, ανισότητα τι κάνουμε. Τι κάνουμε κύριε Καλβέτ. Η ανισότητα, οι ανισότητες καλύτερα, είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρονται και στην έκθεση για την ε, ανάπτυξη του 2017. Οι ανισότητες βεβαίως μας αποσχολούν ιδιαίτερα είναι στο επίκεντρο των συστάσεων που κάνουμε προς τα κράτη-μέλη. Πάντα τις αναφέρουμε. Αναφέρουμε πάντα και αυτό το στόχο. Ξέρετε ότι υπάρχουν και μελέτες του ΩΣΑ και άλλες που τονίζουν ακριβώς την ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Είναι και, αίμα, και θέμα ηθικό και θέμα κοινωνικό. Αλλά όχι μόνο. Γιατί με βάση ο καθένας τις αρμοδιότητές του πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Που είναι και οικονομικό πρόβλημα. Γιατί στην ουσία είναι φραγμός στην ανάπτυξη. Άρα πάντα θα είναι μέλημά μας πολέμηση των ανισοτήτων. Επαραλαμβάνω ότι το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό. Το παρακολουθούμε πολύ στενά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βεβαίως, ήδη αναφέρθηκα στην ε, άνηση μεταχείριση που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι να μην μπορούν να παρακολουθούν ε, τις διάφορες εκπαιδεύσεις και καταρτήσεις αυτοί που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν τις ε, εγκύκλες σπουδές και δεν μπορούν τελικά κατόπιν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά, τα έχουμε υπόψη. Αλλά βεβαίω ο καθένα πρέπει να αναλαμβάνει τι ευθύνε του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Έχουμε και εμεί ευθύνε και φυσικά θα τι αναλάβουμε. Βεβαίω όλα αυτά τα λέμε για να υπάρχει μια κάποια συνέπεια στη δράση μας στον κοινωνικό τομέα, αλλά για να επιτύχουμε και περισσότερη ανάπτυξη, απασχόληση και σωστές σχέσεις μεταξύ των γενεών. Για το βαθμολόγιο λοιπόν, θα είναι ένα πολύ χειροπιαστό εργαλείο για να δούμε πώς εφαρμόζονται οι αρχές μας. Και με έναν τρόπο διαφανή όλοι θα μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για μελλοντικές ανάγκες. Οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες θα την χάνουν της ίδιας προσοχής. Ναι, ακριβώς γιατί θέλουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, ε, ώστε οικονομική και η κοινωνική πρόοδος να συμβαδίσουν. Αυτό είναι για μας ε, ο στόχος για τις κοινωνικές και οικονομικές ε, συνθήκες. Και αν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Στο πακέτο που τώρα επεξεργαζόμαστε δεν έχουμε προβλέψει πρόστιμα και με την υπάρχουσα νομοθεσία θα πρέπει λιγάκι να παραμείνουμε σε όσα προβλέπουν ε, οι κανόνες μας. Μιλάμε για δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιολογούν εκείνα το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε την ίδια προσοχή στα κοινωνικά στοιχεία του κοινωνικού πυλώνα Απλώ θέλουμε μια τέτοια προσέγγιση που να εξασφαλίζει ότι εντό του εξαμήνου δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα και τι κοινωνικέ υποθέσει για την ανέχεια, για τη φτώχεια ε, και τη σχετική μα πολιτική. Σε με την κοινωνική ασφάλιση. Βεβαίω αυτό είναι στα χέρια των ε, κρατών μελών, στι εθνικέ αρχέ και αυτό το εκφράζουν και οι νομοθετικέ μα πρωτοβουλίε, αλλά στι διαδικασίε συντονισμού έχουμε ήδη προτείνει τροπολογία με την ε, ενοποίηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Και βεβαίως δεν μπορεί το κάθε εκατός μέλος να έχει τελείω διαφορετικού κανόνες Θα ακολουθούμε τους ίδιους γενικούς κανόνες απλώς τα κάθε μελη μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα ε, έχουν πρόσβαση σε ποια κοινωνικά δικαιώματα, όπως λένε και οι κανόνε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει πάντως να καταπολεμήσουμε τον κίνδυνο της φτώχειας γενικώ βάσει και των στόχων του 2020. Αποφασίσαμε να μην ε, ε, μειώσουμε το επίπεδο φιλοδοξιών μας και με την οικονομική κρίση είδαμε κάποια πράγματα να υποβαθμίζονται και εμεί λυπούμαστε γι' αυτό όπως και εσείς. Όμως ε, στον κοινωνικό πυλώνα έχουμε σαφείς αρχές για την καταπολέμηση της ανέχειας, της φτώχειας. Είναι σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού πυλώνα. Ο κάθε πολίτη θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα ελάχιστο εισόδημα, αυτό είναι μία από τις βασικές μας αρχές. Ο καθένα θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει έναν αξιοπρεπή βίο, με επαρκές εισόδημα, για να το πετυχαίνει αυτό. Θα πρέπει επίσης να προσφέρονται ανάλογε υπηρεσίε. και όσοι βρίσκονται σε ηλικία να εργαστούν θα πρέπει να έχουν την βεβαιότητα ότι μπορούν να βρουν δουλειά. Η αγορά εργασία θα πρέπει να προσφέρει ποιοτικέ θέσει εργασία και να καταβάλουμε εθνικέ και ευρωπαϊκέ προσπάθειε για αυτόν τον σκοπό. Επίση, θα πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά υπέρ τη ε, δραστηρία και ενεργή συμπερίληψη. Έχουμε τα ανάλογα ταμεία που μπορούν να μας στηρίξουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο για την Κοινωνική Ένταξη. Έχουμε ένα φάσμα από εργαλείων στη διάθεσή μας, ένα ολοκληρό πλωστάσιο που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε με όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Ρωτήσατε τι κάνουμε για τις δεξιότητες για την πράσινη οικονομία και την κυκλική. Εδώ η πράσινη οικονομία, όπως και άλλοι τομείς, είναι το μίσο που πρέπει να ε, συμπαρασύρουμε στην προσπαθία μας επιχειρήσεις και εταιρείε. Αυτούς που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας και αυτούς που ζητούν από τους άνθρωπους να εργαστούν. Πρέπει να δούμε τι χρειάζεται η αγορά εργασίας Είπατε ότι κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και χρησιμοποιούμε διαφορετική διατύπωση. Ναι, σίγουρα χρησιμοποιούμε και διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά λόγια. Αυτή είναι και η ομορφιά της Ευρώπης. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα από όλα αυτά, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια αγορά είναι και ένας χώρος όπου οι πολίτες έχουν ανάγκη να αισθάνονται προστατευμένοι. Γι' αυτό καλό είναι η Ευρώπη να βασίζεται στα σημεία συγκλήσεις και συμφωνίας. Εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κοινού και όχι κάθε χώρα μόνη της. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και στο μέλλον στην Επιτροπή. Πάντως πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ δυνατότεροι και θα έχουμε δυνατότερη φωνή και στον εξωκόσμο. Θα μπορούμε να προσπιστούμε τις αξίες μας και τον τρόπο που έχουμε οικοδομήσει αυτή την αγορά εργασίας και την κοινωνία μας, εάν ακριβώς έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας σε επίπεδο ευρωπαϊκό μαζί με τα κράτη-μέλη. Έχουμε μια αγορά εργασία με σκοπό να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη και θέσει εργασία και να μπορέσουν οι κοινωνικοί πολιτικοί και η οικονομική πολιτική να συμβαδίσουν. Χρειάζονται κάποιες ε, νέε ιδέε για το μέλλον τη Ευρώπη. Η συζήτηση είναι ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, αλλά αν θέλετε τη δική μου γνώμη, νομίζω ότι αν εργαστούμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε καλά αποτελέσματα για όλους. ο ιδιαίτερος για αυτού που δυσκολεύονται. Επτά συναλφοί έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Ε, ο κ. Ζολά θα συνεχίσει να προεδρεύει ε, τη συζήτηση και θα δώσει το λόγο στους ομιλητές. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκίον Παλάς. Γκίον, πού βρίσκεσαι. Θα είμαι σύντομος, αλλά δεν θα... Δεν θα μπορέσω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ε, εσκαλώς όμως θα σας δω ε, Να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα. Η ελεύθερη κυκλοφορία ε, προσώπων και εμπορευμάτων υφίσταται, όμως δεν υπάρχει μια πραγματική κοινωνική Ευρώπη, διότι υπάρχουν πολλά κοινωνικά μοντέλα στην Ευρώπη που δεν είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί ανταγωνισμό και τριβές, μια μειοψηφική ένα αλλά ισχυρή αντίδραση στην Ευρώπη και στο έργο της Κομισιόν με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρόλο που δεν εισακουστήκαμε πλήρως βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή να ε, αντιμετωπίσει το θέμα της ε, έλψης ενός κοινωνικού συντονισμού, μιας κοινωνικής εναρμόνισης. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε, να εξισορροπήσουμε την οικονομική με την κοινωνική Ευρώπη. Η ερώτηση όμως είναι πιο συγκεκριμένη. Έχετε την πρόθεση αυτές οι προτάσεις για τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ε, δήλωσης, κοινής δήλωσης Κομισιών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος αυτής της κίνησης, τι θέλετε να επιτύχετε. Χρειαζόμαστε ένα ανώτερο κοινωνικό ε, επίπεδο νομοθεσίας ε, δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλετε να πείσετε τα κράτη-μέλη που διαφωνούν αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Merci. Αλεξάνδρ. Χαίρομαι για τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός ε, τροφοδοτούνται ακριβώς από την έλλειψη μιας κοινωνικής Ευρώπης. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινή αγορά, έχουμε προχωρήσει σε ένα αριθμό πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως όχι αρκετά στο κοινωνικό πεδίο. Αυτά που ανακοινώσατε είναι σημαντικά λοιπόν και θα αποδείξουν στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για αυτούς, για τα δικαιώματά τους και ελπίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό που δημιουργείται στο κοινωνικό επίπεδο και δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη, να τα ενθαρρύνουμε, να κάνουν πρόοδο. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας ακολουθήσουμε. Θα κάνουμε προτάσεις και θα δώσουμε όθηση. Πώς όμως θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιφυλάξεις εκ μέρους των κρατών μελών. Επίσης χαίρομαι για τις ε, προτάσεις που κάνετε, που ενδιαφέρεστε εν πάση περιπτώσει για τις, καινούριους, για τις καινούριες μορφές εργασίας, την ψηφιακή ε, αγορά, ε, με τις διαβουλεύσεις, κοινωνικούς εταίρους κλπ. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Για αυτά τα θέματα επίσης θα κάνετε μια συλλογή δεδομένων, μια καταγραφή της κατάστασης. Γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από έλλειψη πληροφόρησης. Και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και για τους ε, κανόνες που εφαρμόζονται στις ε, συμβάσεις εργασίας. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Τέλος, και δεν θα το αναπτύξω, να σας υπογραμμίσω το εξής. Έχουμε τις παραμεθόριες περιοχές. Τα διάφορα μέτρα που προτείνεται, για παράδειγμα συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, ε, ψηφιακή αγορά, αποσπασμένοι εργαζόμενοι κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα επηρεάζουν άμεσα τις παραμεθόριες περιοχές. Έχετε προβλέψει κάτι το ιδιαίτερο για αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ. Ο κ. Ροσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκη, ευχαριστώ κ. Τάισεν. Οι 20 προτεραιότητες σας είναι πολύ σημαντικές. Μας βρίσκουν σύμφωνους. Και αν κάτι πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε καθυστερήσει. Όμως το ερώτημα στο μυαλό όλων μας είναι τι θα αλλάξει τώρα που τις ανακοινώσατε αυτές οι 20 προτεραιότητες, τώρα που επικυρώθηκαν από τα τρία θεσμικά όργανα κλπ. Και δεν σας επικρίνουμε, είμαστε δίπλα σας, αλλά βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μια μεριά δεν είχαμε ασχοληθεί με πολύ με αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά θέματα τα τελευταία χρόνια. Πιο πολύ ασχοληθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μας ρωτούσαν οι πολίτες μας γιατί δεν ασχολούμαστε. Τώρα ασχολούμαστε. Το ερώτημα όμως είναι αν σε δύο-τρία χρόνια θα έχουμε δει πρόοδο. Σε όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε κοινωνικά δικαιώματα κλπ. Και αν πρέπει να επικρίνω κάτι, μια έλλειψη, είναι η εξής ο δημογραφικός παράγοντας για το μέλλον. Όλη αυτή η εργασία βασίζεται στην κρίση την, την οποία διερχόμαστε τα τελευταία δέκα χρόνια και την οποία δεν έχουμε πλήρως ξεπεράσει. Μια άγρια παγκοσμιοποίηση κλπ. Ε, και τοποθετούμαστε επί αυτό. Όμω, από την άλλη μεριά, για το δημογραφικό πρόβλημα και τη γύρανση του πληθυσμού δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε, δεν έχουμε αρκετά μέτρα. Όμω, τα επόμενα μέτρα, πολλά από αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα μπορεί ε, να αμφισβητηθούν και να υποσκαφθούν από το δημογραφικό παράγοντα. Ε, φοβάμαι ότι θα δούμε φτώχεια στο, στις ηλικίε. Και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί αλληλεγγύη. Και δεν βλέπω στο κείμενό σας πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, συντάξεις. Ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συνδυάσουμε ε, ταυτόχρονα εργασία και σύνταξη. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Ε, προφανώς υπάρχουν και άλλου τύπου προτάσεις που θα πρέπει να εξετάσετε. Σοφία Ριμπέριο. Κυρία Επίτροπη, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, ήθελα πρώτα απ' όλα να παρατηρήσω ότι βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια τη θητεία αυτή υπάρχει πραγματικά μια εξέλιξη μεταξύ τη ισορροπία μεταξύ τη κοινωνική διάσταση από τη μία και τη οικονομική από την άλλη. Το βλέπουμε από τη δουλειά σα και, και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επειδή το ΕΛΚ αγωνίστηκε πολύ για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία και το λέω ω εισηγήτρια, τέλο πάντων και εισηγήτρια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τα θέματα των κοινωνικών ε, ζητημάτων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όταν μιλάτε για νέου δείκτε ε, στα κοινωνικά ζητήματα για όλε τι χώρε, αυτό είναι σημαντικό ακριβώ και ω προ την πρωτοβουλία για να επιβεβαιώσουμε ξανά την ανάγκη να αμβληθούν οι ανισότητε. Ωστόσο, η άμβληση αυτών των ανισοτήτων θα πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με συγκεκριμένε διαδικασίε ώστε οι χώρε, τα κράτη-μέλη, να ε, εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένε ανισότητε. Αυτό για να πετύχουμε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και ακριβώ να περάσουμε στον κοινωνικό πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος πρέπει να επανασταθμιστεί. Εδώ έχω κάποιες ε, αμφιβολίες σήμερα. Δεν κατάλαβα πολύ καλά και το ομολογώ πώς θα γίνει η διάρθρωση μεταξύ αυτής της νέας πρότασης που την καλωσορίζουμε φυσικά, θέλουμε ένα κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα συζητούμε και διαφορετικά επίπεδα ευρωπαϊκής ολοκλήρωση και ενταξή με τη λευκή βίβλο που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μου φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε ε, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα κοινωνικής ολοκλήρω... Ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως προτείνεται με τα πέντε σενάρια που αναφέρονται στη Λευκή Βιβλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω από τη δική σα την οπτική γωνία Πώς θα γίνει αυτή η διάρθρωση μεταξύ των όσων ζητημάτων εγείρει η Λευκή Βίβλος και η τόσο φιλόδοξη πρόταση για τον κοινωνικό πυλώνα. Και επίση θέλω να επιθέσω την προσοχή πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, σε δύο θέματα. Πρώτον, την ανάγκη να προλάβουμε τις προκλήσεις και τα μελλοντικά προβλήματα συντονιζόμενοι σε επίπεδο θεσμικών οργάνων ε, αλλά και στο επίπεδο των επιχειρήσεων και τη εκπαίδευση, ώστε να υπάρχουν ψηφιακέ δεξιότητε και οι ανάγκε τη τεχνητή αφήγηση να καλύπτονται για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση δεν είναι δική μα αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια διάρτωση με τι ανάγκε των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουμε να προάγουμε αυτέ τι νέε δεξιότητε που περιγράφησαν και να δούμε και την κοινωνική οικονομία. Μια πολύ ε, σημαντική ε, διάσταση που αφορά 2.000 επιχειρήσεις και 14.000 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να έχουμε ένα κοινό ορισμό και να δούμε ακριβώς τι εννοούμε με την κοινωνική οικονομία, με τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτά θα πρέπει να οριστούν με, με, ένα, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει ένας ευρωπαϊκό ορισμός για την κοινωνική οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Μωρά Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μας δώσατε μία νέα πνοή γιατί καταστήσατε σαφή τη βούλησή σας για να υπάρξει μία κοινωνική Ευρώπη. Αυτή η βούληση έγινε κατανοητή από όλους τους συμπολίτες μας. Θέλω να επιμείνω όμως επί του εξής πρωταρχικού. Βεβαίω πρέπει να καταστεί σαφέ ότι μια κοινωνική Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει δυναμική οικονομική αύξηση και αύξηση τη απασχόληση. Αυτή η σχέση μεταξύ μιας δυναμικής οικονομίας και της κοινωνικής προστασίας πρέπει να καταστεί σαφή διότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κοινωνική κατάσταση εξ νύχυλο, εάν δεν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν ε, παρερμηνίες από αυτού του θέματος. Δεύτερον, επί του οποίου θέλω να επιμείνω, είναι οι νέοι τύποι εργασίας, που σχετίζεται ακριβώς και με την ε, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Πρέπει να καταστεί σαφές λοιπόν ότι τα επαγγέλματα που μας παρήχαν τη μεγαλύτερη απασχόληση πριν από 10 χρόνια τώρα έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει τρομερή διακύμανση στα είδη εργασία που προκύπτουν. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει η κατάρτιση. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και στατικά τα προγράμματα κατάρτισης γιατί αλλάζει συνεχώς η κατάσταση. Πρέπει στην ουσία απλώς να χορηγούμε δεξιότητες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες ε, κατηγορίες επαγγελμάτων. Όπως είπατε και εσείς ε, πολύ σωστά κύριε Επίτροπε προηγουμένως, ούτως ώστε να αξιοποιείται και η πείρα στην απασχόληση, ούτως ώστε τελικά κανείς να μην αποκλείεται. Βεβαίως διαβίου κατάρτιση, να ενισχύουμε τις δεξιότητες, αλλά να βασιζόμαστε σε είδη κατάρτισης που να μπορούν να βοηθήσουν για πολλά είδη επαγγελμάτων. Και κάτι άλλο που ήταν πολύ σαφές και στην ανακοίνωσή σας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η αποφασιστικότητα. Ε, αν δεν επιδείξουμε και με βλέπει και η Αγνιές Γιουγκέριους με την οποία συνεργαστήκαμε και για την ε, αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την απόσπαση. Αν δεν υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση και τρομερή επιμονή για να επιτύχουμε, δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, ότι είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα και ναι, πρέπει να κάνουμε πολύ δρόμο για να το επιτύχουμε, αλλά πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε ξενοφοβία και άνοδο των εθνικισμών. Πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Είναι θεμελιώδης. Και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πήγαινε προς διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τις προσπάθειές μας για τους ε, αποσπασμένους. Ιδιαίτερα για τις εταιρείες τύπου Ryanair που έχουν ε, την τάση ακριβώς να κάνουν ε, κοινωνικό dumping. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Η κυρία Ροντρίγιος. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, βεβαίως, το 2017 πρέπει να είναι βασική χρονιά για να αναπτυχθεί η κοινωνική Ευρώπη. Όπως βλέπετε εδώ στην Επιτροπή μας, χαιρετίζουμε την πρότασή σας. Να γίνει μια διακήρυξη για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Οι δύο αρχές που μας προτείνετε, βεβαίως, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίως, αντανακλούν και την έκθεση του Κοινοβουλίου. Αλλά το βασικό μας μέλημα είναι να εφαρμόζονται αυτά που αποφασίζουμε. Ο κοινωνικός πυλώνας Α, πρέπει να υπάρχει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ε, Ευρωζώνη. Στόχος μας πρέπει να είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τον τύπο εργασίας, θα πρέπει να έχουν μια σαφή και αξιοπρεπή σύμβαση εργασίας και να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Χαιρόμεθα που ξεκινήσατε διαβολευούμενοι με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά εμείς θεωρούμε ότι ναι μεν ελπίζουμε να βοηθήσουν οι κοινωνικοί εταίροι για να υπάρξει συμφωνία, αλλά αν δεν βοηθήσουν τότε θεωρούμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να είναι διατεθειμένη να προτείνει νομοθέτημα. Τώρα όμως, να ασχοληθώ κυρίως με την Ευρωζώνη Κοιτάξτε, θα μιλήσω ανοιχτά. Το πακέτο στην τωρινή του κατάσταση, καθώς και το έγγραφο συζήτησης, δεν πηγαίνουν στο βάθος που θα θέλαμε. Και ξέρω ότι εκπονείται και ένα έγγραφο για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τι εννοώ λοιπόν. Αν θέλετε να υπάρξει στην Ευρωζώνη οικονομική και κοινωνική, και κοινωνική συνοχή προς τα πάνω, πρέπει να έχουμε και κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και να ε, μας απασχολεί και η αλληλεπίδρασή τους. Τι εννοώ δηλαδή. Πρέπει να έχουμε μία διαδικασία, μέσω της οποίας για να αυξηθούν οι μισθοί θα πρέπει να αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα για να υπάρξει αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων θα πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με τις ε, εισφορές και την φορολογία. Για να υπάρξει περισσότερη κινητικότητα πρέπει να υπάρχει ε, συντονισμός προς το καλύτερο των κανόνων για τις επενδύσεις. Μόνο έτσι θα έχουμε πραγματική ουσιαστική οικονομική και κοινωνική σύγκληση στην Ευρωζώνη. Και αυτό ακριβώς θέλω να επιτευχθεί. Οι αρχές αυτές αναφέρονται, πρέπει να αναφέρονται σαφώς σε αυτό το έγγραφο που εκπονείται για την Ευρωζώνη. Για να, για να υπάρχει αυτή η σύγκληση προς τα πάνω, στην πράξη, στην πραγματικότητα, να είναι γνήσια, πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και άλλα, αλλά πρέπει να υπάρξει και αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να βασίζεται σε μια δημοσιονομική ικανότητα. Το πακέτο λοιπόν που μας προτείνατε είναι πολύ σημαντικό για τον κοινωνικό πυλώνα, αλλά δεν επαρκεί. Πρέπει τα κοινωνικά θέματα να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και στα επόμενα κείμενά σας, ιδιαίτερα αυτό για την ΟΝΕ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και όλα όσα είπατε σε σχέση με τον κοινωνικό πυλώνα στην Ευρώπη. Στηρίζω προφανώς τον στόχο μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Το ερώτημα είναι πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη. Εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση στην αγορά εργασίας που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συνεπώς μια ενιαία προσέγγιση δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Πάρτε παράδειγμα την Ισπανία. Πολύ ψηλό δίκτυο ανεργία. Αν θέλουμε να επενδύσουμε σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους, δεδομένου ότι οι πόροι δεν είναι πάρα πολλοί, θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί και να εξασφαλίσουμε μια ευελιξία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους ανάγκες. Πώς λοιπόν η Κομισιόν θα λάβει υπόψη αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να προταθεί από την Κομισιόν να υφίστανται ελάχιστε απαιτήσει. Επίση για την ισορροπία μεταξύ του επαγγελματικού και προσωπικού βίου, τι πιστεύετε. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαρτά. Όταν μια επιχείρηση κλείνει επειδή πουλάει προϊόντα που δεν βρίσκουν πελάτες γιατί ε, έχουν παλιώσει, είναι κακής ποιότητας κλπ. Είναι δραματικό, αλλά τουλάχιστον το καταλαβαίνουμε σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό που είναι δραματικό είναι όταν οι επιχείρησει μας κλείνουν όχι επειδή δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, αλλά επειδή μετακινούνται σε χώρες που διαθέτουν ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, ε, ε, όπου ε, απαλλάσσονται από φόρους, όπου το εργατικό δυναμικό είναι πολύ φτηνότερο και πολύ συχνά χάρη σε ευρωπαϊκές για παράδειγμα την Πολωνία. Το σύνολο τη Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής που εισπράττει η Πολωνία ε, ισοδυναμεί με το 3% του ΑΕΠ της. Χωρίς αυτές τις ευρωπαϊκές ε, χωρίς αυτή την ευρωπαϊκή βοήθεια, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την Πολωνία οικονομικά να δημιουργήσει τέτοιου είδου ζώνε. Αυτέ οι επιχειρήσει, οι οποίε λοιπόν απαλλάσσονται και εγκαθιστώνται εκεί, μπορούν επίση να λάβουν να συμμετάσχουν στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνεπώς να πρημοδοτηθούν διπλά. Μιλώ για την Ούλπουλ. Ε, θέμα πολύ σοβαρό στη Γαλλία. Αλλά δεν είναι η μόνη η Whirlpool. Η μόνη τέτοια επιχείρηση και σίγουρα υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις και εκτός της Γαλλίας. Αυτές οι μετακινήσεις δεν είναι αθέμητες. Δεν ε, κινεζοποιούν την οικονομία μας. Δεν ενισχύουν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και πώς σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους μετακινήσεις, αθέμητες μετακινήσεις επιχειρήσεων. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, οι ενισχύσεις τελειώνουν το 2022. Αν λοιπόν δεν, αν σταματήσουν, αυτές οι επιχειρήσεις θα φύγουν και από την Ευρώπη. Θα πάνε στην Ασία και στην Ινδία. Τα ευρωπαϊκά ταμεία λοιπόν μήπως βοηθούν αυτές τις πολυεθνικές εταιρείε να μαζέψουν λεφτά έτσι ώστε τελικά να μετακινηθούν εκτός της Ευρώπης και να μας πουλούν μετά, πουλούν μετά τα προϊόντα τους ακόμα πιο φτηνά. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινωνικό πλεόνα, πολύ σωστά, απόλυτα σύμφωνος, αλλά Είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική αν η Ευρώπη δεν διαθέτει ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Συνεπώς τα πράγματα με τη σειρά τους. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και να αποφύγουμε τέτοιου τύπου αθέμητο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Λέω και Ζόλα πολλές οι ερωτήσεις όπως βλέπετε, εκφράζονται όλα, όλες οι απόψεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο καταρχήν. Uh, okay, honorable uh, members. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις, για αυτά τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω ένα προς ένα. Καταρχήν, ο στόχος και η φύση του κοινωνικού πυλώνα. Ο στόχος, όπως έχουμε πει, είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική σύγκληση, τις αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας που θα πρέπει να είναι πιο προετοιμασμένα εναντί ενδεχόμενων κοινωνικών ε, οικονομικών κραδασμών. Επίσης θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές στην κοινωνία και στον τρόπο εργασίας, τις μορφές εργασίας που αποτελούν το χαρακτηριστικό της κοινωνικής οικονομίας αγοράς του 21ου αιώνα. Επίσης το έγγραφο αυτό θέλουμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς, πλαίσιο για τη δράση των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος λοιπόν είναι μια κοινή ε, δήλωση, διακήρυξη των τριών θεσμικών οργανών. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το καταφέρουμε, αλλιώς ο πυλώνας θα παραμείνει σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τον προβάλαμε αρχικά. Μετά, για τη σχέση ανάμεσα στον πυλώνα και την Λευκή Βίβλο. Την ίδια ακριβώς μέρα που παρουσιάσαμε τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, δημοσιεύσαμε και ένα έγγραφο ε, για ε, την κοινωνική Ευρώπη, μια λευκή βίβλο ε, δηλαδή. Ο πυλώνας είναι η πρόταση της Κομισιόν για την ενίσχυση της πολιτικής προσήλωσης σε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση Ευρώπης. Το έγγραφο περί είναι πιο μακροπρόθεσμο, έχει πιο ευρύ ορίζοντα, πώς μπορεί δηλαδή, να, ποιες είναι οι εξελίξεις που μπορούμε να προβλέψουμε, οι τάσεις και μέσω αυτού εξετάζουμε τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου για το κοινωνικό κεκτημένο. Έτσι συνδέονται οι διάφορε πρωτοβουλίε στα διάφορα έγγραφά μας, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, συνοδευτικές πρωτοβουλίες Γι' αυτό το θέμα έχω να σας επαναλάβω ότι θα ξεκινήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους μια διαβούλευση η οποία όμως ακόμα και αν δεν καταλήξει κάπου δεν σημαίνει ότι δεν θα υποβάλουμε προτάσεις. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που έγινε με το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον προσωπικό βίο. Μετά, για το ζήτημα των δημογραφικών εξελίξεων και το πώς τις πήραμε υπόψη στον κοινωνικό πυλώνα. Όταν αναπτύσσουμε δικαιώματα και αρχές στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τις δημογραφικές εξελίξεις. Χρειαζόμαστε βιώσιμα, διατηρήσιμα κοινωνικά συστήματα και ασφαλώς το δημογραφικό έχει ληφθεί υπόψη. Πιο πολύ όμως στο έγγραφο εργασίας για την κοινωνική διάσταση που είναι και πιο πακροπρόθεσμο. Μετά ε, υπόθηκε ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τις κοινωνικές με τις οικονομικές τυχές της Ευρώπης. Το έχουμε προσπαθήσει στο έγγραφό μας. Δεν πρόκειται να πετύχουμε την κοινωνική σύγκληση χωρίς να πετύχουμε και την οικονομική σύγκληση. Άλλωστε, η οικονομική σύγκληση θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε και σε πολλά άλλα προβλήματα που δημιουργούνται, όπως η αθέμητο, ο αθέμητος ανταγωνισμός, οι ε, αποσπάσεις εργαζομένων κλπ κοινωνική και οικονομική σύγκληση θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Κατόπιν, το θέμα των δεξιοτήτων. Το είπα και στην πρώτη μου απάντηση. Οι δεξιότητες είναι τμήμα της απάντησης που θα πρέπει να δώσουμε. Θα παραμείνουν σημαντική προτεραιότητα της Κομισιόν. Το θέμα τώρα το, του κατά πόσο ο κοινωνικό πυλώνα αφορά την Ευρώπη ή τη ζώνη του ευρώ. Αυτή τη στιγμή έτσι όπω το έχουμε, τον έχουμε προτείνει αφορά όλη την Ευρώπη αλλά σχεδιάστηκε κυρίω για τη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή είναι ανοιχτό ο κοινωνικό πυλώνα για όλη την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο ότι σχεδιάστηκε για την ζώνη του ευρώ. Κατόπιν, δημοσιονομικές δυνατότητες. Εδώ είναι ένας τομέας στον, για τον οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο για την ε, ε, ε ολοκλήρωση της ε, οικονομική και κοινωνική Ευρώπης ε, που θα υποβάλουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Θα πρέπει λοιπόν όταν ε, ολοκληρώσουμε την, ε, στο έγγραφο για την ολοκλήρωση τη Οικονομικής και Νομισματική Ένωση. συγγνώμη. επίσης μιλούμε για τα, τους συγκρατικούς κανόνες, τα benchmark, ε, για τη σύγκληση Χρειαζόμαστε τέτοιου είδου συγκριτικές ε, ε, ε βαθμολογίες ε, προκειμένου να προχωρήσουμε στην σύνδεση. Τώρα, ελάχιστες απαιτήσει. Αυτά που προτείνουμε είναι ήδη ελάχιστες απαιτήσει. Τα κράτη-μέλη μπορούν να τις υπερβούν. και μάλιστα έχουμε εξετάσει και, και τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και αρνητικό αντίκτυπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ταμεία, τα ταμεία εκ του κανονισμού τους δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούν ε, μετα, αθέμητες μετακινήσεις επιχειρήσεων. Έτσι κι αλλιώς, όταν μιλάμε για κοινωνική σύγκληση, όλοι κατανοούμε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί και η οικονομική σύγκληση και τα ταμεία αυτά, τα ευρωπαϊκά ταμεία, υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την οικονομική σύγκληση. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να διακοπούν οι οικονομικές ενισχύσεις μετά το τέλος του, δημοσιονομικού, του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Διότι τα ταμεία αυτά πραγματικά εξασφαλίζουν την οικονομική σύγκληση. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Τάισον. Για να έχει, θα λέγαμε, την τελευταία λέξη σε όλη αυτή τη συζήτηση για σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να δω τι μπορώ να προσθέσω, γιατί οι απαντήσεις του Βάλντης ήταν ε, πληρέστατες. Βεβαίως ο κοινωνικός πυλώνας αφορά την σύγκληση. Τη σύγκληση όπως είπε μόλις τώρα ο Βάλντης. Και για τις ερωτήσεις των συναδέλφων Μπαλάς και Σαντέρ, Βεβαίω δεν έχουμε ακόμη αρκετή κοινωνική Ευρώπη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζει η κατάσταση και έχουμε νέες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και στα κοινωνικό τομέα λόγω των δημογραφικών εξελίξεων, της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και άλλα μεταβαλλόμενα στοιχεία και βεβαίω η κοινωνική διάσταση πρέπει να ακολουθεί και να βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι κοινωνικές προκλήσεις καλύπτονται. Δεν είναι δικό μας Βεβαίω το καθήκον να τα καλύψουμε όλα, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε σε συνεργασία με τα κατημέλη ότι νέοι ναι, κίνδυνοι καλύπτονται και ότι τους αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως, δεν νομίζω ότι πηγαίνουμε πολύ μακριά, διότι αν δείτε τι καταφέραμε τα τελευταία 60 χρόνια με τις ίδιες ευκαιρίες λόγω χάρη ανδρών γυναικών, είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι, πραγματικά υπήρξαμε πρωτοπόροι και αν δεν είχαμε τότε εκείνες τις πρωτοβουλίες από το ευρωπαϊκό μέτωπο, για να το πω έτσι, ε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε σήμερα. Βεβαίως, δεν έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας ως τώρα, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε πετύχει ως τώρα και τι κάναμε και μας. Με τα 60-70 νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για κοινωνικές υποθέσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν κάναμε και τίποτα για, κοινωνικέ, για τα κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε ένα ολόκληρο κοινωνικό κεκτημένο πίσω μας. Και τα ταμεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να πω και το μικρά κοινωνικά ταμεία της παγκοσμιοποίησης δεν είναι και τόσο ασήμαντο. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε τις μετακινήσεις εταιριών ή την αναδιαρθωσή τους. Ή το ΦΕΑΤ και άλλα ταμεία εάν ε, σκεφτείτε, είναι το 1 δέκατο του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να βοηθήσουν τη στήριξη των κρατών κάποιων συγκεκριμένων περιοχών, περιφερειών και με κοινωνικές επενδύσεις και ούτω καθεξής. Και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βλέπουμε μια ολένα και μεγαλύτερη προβολή στα κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε τη σχετική στρατηγική και τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης. Φαίνονται ε, ήπιοι ως μέτρα αλλά νομίζω ότι τα κάτι μέλη τουλάχιστον μπορούν να διδαχθούν εμένα από του δε. Μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη μέθοδο συντονισμού. Και όλα αυτά μπορούν πραγματικά να είναι υποφελή και να μα ε, βοηθήσουν και στο σχεδιασμό μελλοντική πολιτική. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και μην ξεχνάμε και τι δεξιότητε, ήδη τα είπαμε. Για τον κοινωνικό πυλώνα. Η επίσημη εξαγγελία του Βάλντι ήταν η τέλεια απάντηση ούτω ή άλλω. Αλλά η κοινή εξαγγελία με τα κράτη-μέλη και με τη συμμετοχή του, του Ευρωκοινοβουλίου βεβαίω βοηθά και στην ανάληψη ευθύνη από την πλευρά των εργών μελών. Και με την ανάληψη ευθύνη μπορούμε να προχωρήσουμε και καλύτερα από κοινού. Ελπίζω λοιπόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Και αν όχι, έχουμε τι δικέ μα τι συστάσει και για μα είναι η βάση επί τη οποία θα θεμελιωθεί η μελλοντική μα πολιτική. το τι θα κάνουμε με τις αρχές αυτές στο μέλλον για να δείξουμε ε, ότι αυτό πραγματικά θέλουμε και να υλοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς προβλέψαμε τις τέσσερις συγκεκριμένε δράσεις και θα ε, διαρθρωθεί αυτή η ε, διάθεση να δράσουμε και στα μελλοντικά προγράμματα εργασίας του 18, του 19, όπω έγινε και στο παρελθόν, με αρκετά βήματα συμφωνία και να είμαστε φιλόδοξοι, να είμαστε φιλόδοξοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη θητεία για τα επόμενα δύο χρόνια. Πιστεύω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε και ήδη να έχουμε κάποιε πρώτε προτάσει. Οι δημογραφικέ εξελίξει, όντω, μια από τι βαθύτερε αλλαγέ. Μια από τι αλλαγέ που, πώ να το πω, μα ενθαρρύνει, μα οδηγεί να προχωρήσουμε σε αυτέ τι αλλαγέ. Έχουμε την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιοποίηση, αλλά κυρίω οι δημογραφικέ εξελίξει. Εάν δείτε τις αναχώρασεις τάσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι σημαντικό και πρέπει να δοθεί συνέχεια. Κάτι που πρέπει να πω, πώς να το πω, δεν είναι απλό να σχεδιάζει κανεί πολιτική και με τη μία να δίνει τη σωστή απάντηση σε τέτοιε μεγάλε αλλαγέ. Όμω, εάν κανεί παρατηρεί με προσοχή το τι συμβαίνει τώρα, μπορεί κάπω να ε, σκεφτεί τι θα γίνει σε 20-30 χρόνια. Δεν ξέρουμε πόσου ακριβώ ηλικιωμένου θα έχουμε τότε. Όμω, αν είναι κανεί ξύπνιο, μπορεί να προετοιμαστεί εγκαίρω. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάναμε όταν ζητήσαμε από τα κάτι μέλη να αλλάξουν τα συνταξιδοτικά του συστήματα. Δεν ήταν ο στόχο να κάνουμε μαύρη τη ζωή των ανθρώπων. Ήταν να έχουμε συστήματα τα οποία να είναι βιώσιμα, να αντέξουν στο μέλλον. Και κοιτάμε και το κατά πόσο τα ε, συστήματα αυτά μπορεί να είναι επαρκή, δηλαδή να δίνουν και κάποιε συντάξει εξωπρεπεί όταν φτάσουν ε, στο όριο τη σύνταξη οι άνθρωποι. Το πώς συνδέονται ο κοινωνικός πυλώνας με το έγγραφο ε, μελέτης και αυτό το απάντησε νομίζω ο αντιπρόεδρός μου, ε, οι ψηφιακές δεξιότητες και αυτό τέθηκε ως ερώτηση. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι 90% των μελλοντικών θέσεων εργασία ήδη σήμερα, για να μην πω το μέλλον, απαιτούν ψηφιακέ δεξιότητε. Και είδαμε ότι ένα στου 10 ε, σε ηλικία εργασία δεν τι έχουν αυτέ τι δεξιότητε. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό αναπτύξαμε ως πρώτη προτεραιότητα ε, ε, του καταλόγου για τις ε, δεξιότητες, τις ψηφιακές, για να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να απασχοληθεί και στην αγορά των ψηφιακών θέσεων εργασία. Για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και είδαμε να το στηρίζουν και τα κρατη και το κοινοβούλιο. Και υπάρχει διάθεση να προσφερθεί η δυνατότητα αυτή στου πολίτε να αναπτύξουν τι δεξιότητέ του, τι βασικέ ψηφιακέ δεξιότητε. η οικονομία, περισσότερες ε, διατομεακές δεξιότητες ε, για να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον, συνεργασία με όλους τους εταίρους, ναι, ε, για όσους σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, για τους εργοδότες, τους ενδεχόμενους εργοδότες, τους επιχειρηματίες, τους συνδικαλιστές, τους κοινωνικούς εταίρους και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα μας βοηθήσει εδώ πέρα με τεχνικές που έχουν δοκιμαστεί. Και η Eurostat μπορεί να εξυπηρετήσει με νέες τεχνικές για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες για το μέλλον, τι είδους εκπαιδευτικές ε, δεξιότητες θα χρειαστούν. Και μια παρατήρηση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το τι ε, μπορεί να μας πει για τα θέματα αυτά ο Γενικός Εισαγγελέας. Είναι καλό να υπάρχει ένα τέτοιο ε, διεξοδικό έγγραφο, ένα ενιαίο κείμενο που να εξηγεί το τι ισχύει για την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει νόημα να ανήκει κανείς στο σύστημα ασφάλισης ενός κράτους μέλους με, μια σύμβαση Όμως, το θέμα είναι πώς θα οργανώσουμε εμείς τη σχετική νομοθεσία. Ε, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι αν υπάρξει πρόβλημα πρέπει από κοινού με τα κράτη-μέλη, με τη διοικητική επιτροπή και τη σχετική διαδικασία να το δούμε το, το πρόβλημα. Υπάρχει σχετική διαδικασία και πριν την ε, οδηγία για την ε, εφαρμογή ε, δεν ήταν σαφέ. Η οδηγία εφαρμογή το ξεκαθαρίζει. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να δουλέψουν μαζί. Το ξεκαθαρίζει εδώ και κάποιου μήνε και αν όλα τα κράτη-μέλη παίξουν σωστά το ρόλο του, πιστεύω ότι μπορούμε με αυτή τη διαδικασία να λύσουμε πολλά προβλήματα θα δοθεί συνέχεια και στο μέλλον, αλλά ήδη βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ερμήνευσε το ενιαίο πιστοποιητικό και νομίζω ότι έχουμε πια τις διαδικασίες και απλώ μπορούμε να τι ακολουθούμε. Και τα κάτι μέλη έδειξαν ότι θα συνεργαστούν. Οι οι διαδικασίε προφανώ δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Κάτι άλλο που υπόθηκε ήταν ένα όραμα του Γενικού ε, Εισαγγελέα για την ε, άγρα δικαιοδοσία. Εδώ δεν θα σχολιάσω τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως, το δικαστήριο που θα ασχοληθεί με τα κοινωνικά ζητήματα είναι και αυτό όπου ουσιαστικά θα εδράζονται τα βασικά συμφέροντα του εργαζομένου, ελπίζω. Ε, αλλά θα φανεί και από την τελική απόφαση του δικαστηρίου αυτό. Και συμφωνώ με την κυρία Ροντρίγκε και με αυτά που υποβάλλει ότι βεβαίω το έγγραφο μελέτη, τα έγγραφα μελέτη πρέπει να συνδυαστούν. Είναι ένα σύνολο και όλα εξυπηρετούν το διάλογο και τη συζήτηση, την ευρύτερη για γύρω από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον τη Ευρώπη. Εάν μιλάτε για του διάφορου τομεί και την εμβάθυνση τη συνεργασία, βεβαίω δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να λέμε το ένα είναι κοινωνικό, το άλλο οικονομικό. Όχι, αυτά πηγαίνουν από κοινού, χέρι-χέρι. Και πρέπει να υπάρξει ένα κοινό πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εμπλουτίσουν αυτή τη συζήτηση. Ιδίω ε, όταν ε, πήραμε κάποιε αποφάσει για τα κοινωνικά ζητήματα την περασμένη εβδομάδα, αυτά δεν θα είναι σε ένα στεγανό ξεχωριστά τα υπόλοιπα, αλλά θα το συνδυάσουμε με τα υπόλοιπα. Η παγκοσμιοποίηση, η εμβάθυνση τη Νομισματική Ένωση, όλα αυτά μα ενδιαφέρουν σε συνδυασμό με τα κοινωνικά στοιχεία και πρέπει να ισχύουν παντού. Και για την κυρία Στίβεν, με τελευταία απάντηση. Όταν ε, καταρτίζουμε νομοθεσία στην Ευρώπη, πάντοτε κοιτάζουμε να ζητούμε το ελάχιστο που μπορούμε από τα κράτη-μέλη. Έχουμε κανόνε ελάχιστου. Ε, και τα κράτη-μέλη, εξελαχίστων μάλλον, και τα κράτη-μέλη μπορούν πάντοτε κάτι να προσθέσουν ε, βάσει του άρθρου 53 τη συνθήκη. Αυτό γιατί έτσι, όχι απλώς γιατί έτσι μας αρέσει να είμαστε οργανωμένοι, αλλά γιατί το ορίζει ήδη η συνθήκη. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε όλη εμπιστοσύνη ότι τα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις θα κάνουν μια προσπάθεια να κάνουν και κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας, αλλά κυρίως για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και για τις απαντήσεις. Ο διαφρομένος διάλογος είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημοκρατία μας. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν στοιχείο η παρουσία σας εδώ. Η Επιτροπή με την ενέργεια αυτή δίνει μια ευκαιρία στην κοινωνική Ευρώπη. Από ό,τι ακούσατε από τους συναδέλφους, από την αδημονία ορισμένων εξ αυτών, δείχνει πόσο θέλουν να υπάρξει πρόοδος για το θέμα αυτό, πόσο θέλουν και οι ίδιοι να βάλουν πλάτη. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να απαντήσουμε στις απόλυτα αιτιολογημένες ε, προσδοκίες των πολιτών μας. Αν υπάρχει μια ευχή που θα μπορούσα και εγώ να κάνω για να κλείσουμε αυτή τη ζήτηση, είναι αυτή η ευκαιρία που έχει η κοινωνική Ευρώπη να μην είναι απλώς ε, ένα μικρό βήμα προς τα μπρος, είναι να γίνουν πραγματικά σημαντικά πράγματα. Γιατί ναι, μπορεί εδώ πέρα να υπάρχει αδειμονία αλλά κυρίω υπάρχει στι κοινωνίε μα. Έχετε λοιπόν και έχουμε μια σημαντική ευθύνη για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίασή μα για το επόμενο θέμα που ήταν ε, η ακρόαση του υποψηφίου για τη θέση του επικεφαλής του Ταμείου για την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Δυστυχώς πρέπει να αναβληθεί δεν μπορεί να λάβει χώρα. Οπότε θα τα πούμε αύριο στις 9.30. Θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες απευθείας και ευχαριστώ πολύ.